Άρχεται η συνεδρίαση. Πάμε στην έκθεση Πάσκου. Κύριε Σιγητά, έχετε την δυνατότητα και την ευκαιρία για μια τελευταία παρατήρηση. Comment. σχόλιο. Δεν είμαι ένοχος, αθώος. Ερχόμαστε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Συμβαστική 1, υπέρ. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Άλλη μια φορά. Ποιος είναι υπέρ της 51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 it's closed before. It's been 28 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται, λέει ο πρόεδρος. You have exchanged your cards and all... Αλλάξατε τις κάρτες σας. You, the, you vote all on one card. Όλοι με μία κάρτα ψηφίζετε. Για να είμαστε σίγουροι, ας ξαναψηφίσουμε τη συμβιβαστική τρία. Όχι, την 51. Τροπολογία 51. 51. Ναι. Σάκε, τροπολογία Σάκε. Είστε ουδέτεροι. Η Πέρα τη ψηφοφορία. 28-28. Απορρίπτεται. Άρα απορρίπτεται. Έφυγε ο συνάδελφος πριν την ψηφοφορία. Πάμε τώρα στην 52. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τότε στην τροπολογία 73. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Το δεύτερο τμήμα μάλλον πρώτα. Τι υπάρχει εδώ. Λέμε 51 της, 50, της 73. Εδώ έχει γραφτεί τελείως χαζοδός. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108. Τροπολογία 108. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 λέει ο πρόεδρος. Α, μόλις την ψηφίσαμε. 148-149. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, καταπίπτει μάλλον, καταπίπτει όταν ε, απορριφθεί το δεύτερο τμήμα. Είναι το φαινόμενο ντόμινο. Φτάνουμε τώρα, καταπίπτουν όλα και πάμε στο 153. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται 156. Υπέρ. Δεν πέφτει, δεν καταπέφτει. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 153 λέει ο πρόεδρος. 163 διορθώνει. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ. 164 υπέρ. Κατά αποχές. Μπορείτε να κλείσετε το στόμα σας. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ καταπίπτει. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη 12. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 200. Τροπολογία 300. 200. Πρώτο τμήμα. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στο δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ. Κατά αποχές αλέχουμε. Τη 220. Πέρα στις ψηφοφορίες. Ε, απορρίπτεται. 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 222, 223, 224 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε. Συμβαστική 14. Πέρα της ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα. Πάμε στην συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 256. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ 72 κατά αποχές εγκρίνεται 273 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παρακαλώ 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 275 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι, αυτό καταπίπτει. Επειδή έχουμε εγκρίνει τη 17. 76-77 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 να όχι καταπίπτει πάμε στη συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε Πέρα τη ψηφοφορία. 40 με 19. Εγκρίνεται. 97, 297 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία, συνάδελφοι. αλλιω να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 297 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 299 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη 299. Πέρα στις ψηφοφορίες. 31 προς 28. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 300-301 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε. Πέρα της ψηφοφορία. 26 προς 32 απορρίπτεται. 306 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 307 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 309 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 311 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 312 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 313 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 314 απαράδεκτη μία αποδεκτή τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται προφορική τροπολογία 5 ευχαριστώ Πρέντα. Δεν έχει διαφορά. Ποιο είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Και 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 και 13 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία όλης της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Η της ψηφοφορίας. 36 υπέρ 18 κατά 5 αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Κυρία Λόζινγκ. Έχουμε κατοθήσει μία έκθεση με ψηφίας και τη στείλαμε στην γραμματεία την προηγουμένη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το διεκπαιρεώσουμε. Πάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου ΠΑΤ για την Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλει να πει ο εισηγητής. 91 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τότε στην 103. Αν την βρω. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Εκατόν τρία. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Παρακαλώ. ist doch gut, dass ich manchmal Abstimmung zweimal aufrufe. Äh, damit ist Εγκρίνεται. Είναι καλό που καμιά φορά ψηφίζουμε και έτσι. Έχουμε κάνει μία αποχή, κατά, αποχές. Όχι, ψηφίσατε αποχή. Α, ωραία. Ευτυχώς που μου το είπατε. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. thought it was part three. Νόμιζα ότι ήταν το 3. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε 104. Υπέρ. Κατά. Ανακατοσούρα. Λοιπόν, 104. Γιατί τα πλέξαμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 3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 Κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 138. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. 31 ψήφοι υπέρ, 28 κατά εγκρίνεται, 141 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, 144 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 157 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ζητήσω από τους συναδέλφους από το ΕΛΚ να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία. Πάμε στην 186. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 188-189 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 249 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 250 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 251-52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά αποχές. Άλλη μια φορά. 258 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Πέραστη geschlossen. ψηφοφορία. 24 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Πέρασε τα ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 30 κατά. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην 274-75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 277 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ, κατά αποχές Άλλη μια φορά, 282 υπέρ. Κατά, Ελέγχουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. 23 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 284 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 286 και υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 288 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 287 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 289 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 293, 94, 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 297 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Στροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές. Η 59 για να ελέγξουμε. Το κάνουμε πιο συχνά γιατί είναι πολύ μικρή η συμμετοχή στην ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 25 υπέρ, 18 κατά. Και 15 Αποχές. 25 λοιπόν. Εγκρίνεται. Πάμε στην 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 25. Υπέρ. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και έτσι φτάνουμε στην τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε.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 Πέραση της ψηφοφορίας. 37 ψήφοι υπέρ, 20 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια για την έκθεση. Πάμε τώρα στην έκθεση Λούλατσεκ. Κυρία Λέζινγκ. Yes, Έχουμε καταθέσει μια έκθεση μειοψηφία. Τη στείλαμε στην Γραμματεία την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία. Πάει πολύ καλά. Πάμε τώρα λοιπόν στην έκθεση Λούνατσεκ. Εδώ υπάρχουν τρεις τροπολογίες που είναι όμως ταυτόσιμες και θα τις ψηφίσουμε μαζί. Την 1, 2, 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Was kriege ich, Ulrike? Τι παίρνω, Ulrike? Πέρα τη ψηφοφορία. 45 υπέρ. 5 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. Κάπως αλλιώς ήτανε που το περιμένατε. Ε. Τι συμβαίνει. Ουλρίκε. Ουλρίκε. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς ψηφίζουμε τώρα, συγγνώμη. Ξέρω, αλλά ποιο τμήμα, το πρώτο τμήμα. Την παράγραφο 1, της τροπολογίας 1, 2, 3. Μπενιφέη, Κασπάρη, Κούκαν. Υιοθετήθηκε 45 υπέρ, 11 κατά. Εκτός μικροφώνου κυρία Λουνατσέκ. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σχέδιο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 46 ψήφοι υπέρ 7 κατά 3 αποχές. Κυρία Λούλα Τσέκ. Ναι, τώρα θέλω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αποσύρω την, το όνομά μου από αυτή την νομοδότηση γιατί δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι είναι μισογεμάτο το ποτήρι και να συγκατατεθώ. Ξέρω ότι έγινε πολύ πρόεδρος και γι' αυτό το συνοδευτικό ψήφισμα έχει θετικά στοιχεία. Όμως γι' αυτό εδώ θέλω να αποσύρω το όνομά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Hm? What? agree Δεν συμφωνεί να διαρθώσει την ψηφία Δεν είναι ονομαστική. Είναι ονομαστική. Δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε λοιπόν και πέρα η έκθεση όπως συνήθως στην Ολομέλεια. Είναι η συνήθις διαδικασία. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε τώρα στην έκθεση Λούνατσεκ. Αυτή είναι Λούνατσεκ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρά που δεν την ελληπή συμμετοχή του ΕΛΚ. Έχουμε ανθρώπους από το ΕΛΚ που δεν έχουν ψηφίσει, τα δύο τρίτα. Η παράγραφος 1 θα πρέπει να ελεγχθεί ηλεκτρονικά. Μάλλον η τροπολογία 1 διορθώνει ο πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συ... Τροπολογία πάμε τώρα την 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 20 κατά, 11 αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, γιατί δεν βλέπω χέρια. Πέρα της ψηφοφορίας, 40 υπέρ 13 κατά εγκρίνονται. Πάμε τώρα στην 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 σε τέσσερα τμήματα ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, όχι, ελέγχουμε. Τέταρτο τμήμα, ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίες. 11 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 15 αποχές. 29, δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Υπέρ, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ δεύτερο τμήμα να το ελέγξουμε ωραία πέρα στις ψηφοφορίες 9 υπέρ 31 ψήφι κατά απορρίπτεται είσαι και εσύ λίγο υπεύθυνη Ουλερίκια 30 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. 48 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές εγκρίνεται. Κυρία Λούνατσεκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και ηγητές για την πολύ καλή του συνεργασία καταφέραμε να βάλουμε αρκετά πράγματα στο κείμενο. Δεν συμφωνώ, όπως είπα προηγουμένως, με την τροπολογία 17, όμως υπερψηφίστηκε και θα διατηρήσω το όνομά μου στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί πιστεύω ότι αυτό το ψήφισμα έχει πολλά θετικά τα οποία στηρίζουν την ε, πρόοδο ε, στην καταπολέμηση της υποχρεωτικής εργασίας στο Ουσβεκιστάν. Κοιτάξτε. Όλα αυτά δεν ξέρουμε πώς θα πάνε, αλλά έχουμε πάντοτε την καλή θέληση. Πάμε τώρα στη δική μου γνωμοδότηση, υπέρ, ηλεκτρονικά καλύτερα. Είναι πιο απλό. Υπέρ. Κατά αποχές. Όχι, ηλεκτρονικά, εντάξει. Και πέρα στις ψηφοφορίες, 40 υπέρ, 3 ε, ψήφοι κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται. Τίποτα για τα διάφορα. Όχι. Επόμενη συνεδρίαση 17-18 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.